Good afternoon. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Η Πρόεδρος, παρακαλώ καθίστε. Good afternoon. Σας ξαναλέω καλό σας απόγευμα σε όλες και όλους. Κυρίσω την έναρξη της απογευματινής συνεδριάσεως και με μεγάλη χαρά αρχίζουμε τη συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γιουλιάνη Μπόγνερ Στράους που είναι Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και θα, θα μιλήσει για τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Η Αυστρία, ως γνωρίζετε, ανέλαβε την Προεδρία πήρε τη σκητάλη από τη Βουλγαρία στην πρώτη εβδόμου. Και ε, με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε από εσά, κυρία Υπουργέ, σχετικά με τις προτεραιότητες, το χρονοδιάγραμμα, κάποια πράγματα πολύ σημαντικά για μας, στην Επιτροπή δηλαδή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι βεβαίως θα απαντήσετε και σε όλες τις ερωτήσεις. Η κυρία Στράους έχει υπάρξει ευρωβουλευτής και είναι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες και με τις καλές και κακές συνήθειες του Ευρωκοινοβουλίου. Ως συνήθως θα σας δώσω τον λόγο, θα τον λόγο στην κυρία Υπουργό για την παρουσίαση για 15 περίπου λεπτά και θα συνεχίσουμε με ερωτήσεις και απαντήσεις, σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής ξεκινώντας πρώτα από τους συντονιστές. Έχει το λόγο κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι συντονιστές, αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου πρώτα να υπογραμμίσω ότι ήμουν βουλευτής της Αυστριακής Βουλής. Η κυρία Κέστιγκερ, υπουργό τώρα στην Αυστριακή κυβέρνηση, ήταν ευρωβουλευτή εδώ, την αντικαθιστώ σήμερα. Ήμουν και υπουργό οικογενειακών υποθέσεων στην Αυστρία, εγώ ίδια. Και τώρα, αντικαθιστώντα την κυρία Κέστιγκερ, σα παρουσιάζω τι προτεραιότητε τη Αυστριακή Προεδρία. Σα μεταφέρω δε του θερμού χαιρετισμού τη Ελισάβετ Κέστιγκερ η οποία γέννησε ένα αγοράκι την Κυριακή. Ολόκληρη οικογένεια χέρι άκρας υγείας. Δεν θα σας ευνηδιάσω λέγοντας ότι το κέντρο βάρους της Αυστρικής Προεδρίας στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής για την συζήτηση των νομοθετικών προτάσεων θα είναι για την περίοδο μετά από το 2020 λόγω του θεμελιώδους ρόλου της ενίσχυσης της ε, περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 1 τρίτο συνολικά των κονδυλίων από το 2021 έως 2027 Επομένως, η πολιτική συνοχή είναι από τους θεμελιώδεις τομεί πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνοχή αποτελεί έκφραση της κοινωνία αξιών και της αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Πολυάριθμα έργα και προγράμματα σε όλες τις χώρε μέλη και τις περιφέρειες επιτόπου λαμβάνουν στήριξη. Έτσι γίνεται ορατή και απτή η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ανταποκρίνονται στις ε, τοπικές ανάγκες και στην βάση της ενισχυμένης στόχευσης σε παράγοντες ενίσχυσης της ε, συγκυρίας και της παραγωγής δεξιοτήτων, τα ταμεία μπόρεσαν να μειώσουν, να απαλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης και να υποστηρίξουν όλες τις περιφέρειες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Γνωρίζουμε ότι η διαμόρφωση των συνθήκων πλαισίων για την άσκηση της πολιτικής αυτής έχει σημασία για όλες τις χώρες μέλη και τις περιφέρειες. Υπό την Αυστριακή Προεδρία αναμένουμε πολλές και σημαντικές συμβολές από όλες τις ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων και βεβαίως και εντατικές ε, διαπραγματεύσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου. Μετά από τη διευκρίνηση των ανοιχτών θεμάτων στην αρχή της Προεδρίας μας, έχουμε τον στόχο μετά να στοχεύσουμε στις πτυχές εκείνες που είναι αναγκαίες για την επόμενη γενεά προγραμμάτων προώθησης. Διότι σημαντική καθυστέρηση της έναρξης των προγραμμάτων όπως διαπιστώσαμε τώρα θα πρέπει να αποφευθεί με κάθε τρόπο. Άλλο σημαντικό σημείο στις διαπραγματεύσεις για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλοποίηση των διαδικασιών και ελέγχου των ευρωπαϊκών ε, χρηματοδοτήσεων. Θα πρέπει να εξεταστεί αν οι υποβληθήσεις προτάσεις κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται πως το πράττουν αυτό. Αν όντως όμως οδηγούν σε αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η απλοποίηση είναι κάτι το οποίο ζητούν όλες οι χώρες μέλη και ιδίως για την μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και για την διοίκηση. Εδώ φάνηκε καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι βελτιωμένες συνθήκες πλαίσια για την καταβολή των κονδυλίων και όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να είναι και κεντρικό πολιτικό αίτημα της μεταρρύθμισης αυτής. Πέρα από αυτό θεωρώ ότι με την απλοποίηση για την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων συμβάλλουμε ισχυρά και στην ενίσχυση της επικουρικότητας. Εν προκειμένου, θέλω ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δηλώσω στα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεως και ιδίως προς τους εισηγητές και εισηγήτριες ε, να δηλώσω τη μεγάλη μου ευχαριστία για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει για την απλουστευμένη πολιτική συνοχής που θα είναι για μας σημαντική προσανατολισμή για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Όσο θα γνωρίζετε υπάρχει ήδη στο τεχνικό επίπεδο μεταξύ των εμπειρογνωμόνων μας σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα κοινά στοιχεία, να βολιδοσκοπήσουμε τα βάθη για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Τόχος και σκοπός της Προεδρίας μας είναι στι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο, έστω και αν η πρόοδος αυτή θα εξαρτηθεί βέβαια από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζουμε ότι τα θέματα της σωστής κατανομής των πόρων, της, του επαρκού ε, όγκου των πόρων, των ε, εθνικών συνεισφορών, θα, θα χρειαστούν προθυμία από όλους τους συμμετέχοντες διαπραγματεύσεις, χώρες μέλη και θεσμικά όργανα. Κυρίως από αυτήν την διαθεσιμότητα και την προθυμία θα εξαρτηθεί εάν το, ο φιλόδοξος στόχος που στηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκαιρη συνεννόηση και συμφωνία για το σύνολο του πακέτου. Στο πολιτικό επίπεδο, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, γίνεται ενημέρωση των Υπουργών Συνοχής και προβλέπεται για τα τέλη Νοεμβρίου η ενημέρωση αυτή. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, εκτός από τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων στο επίπεδο του Συμβουλίου, επιθυμούμε να επιτύχουμε συνέχεια και στις διακρατικές διαδικασίες για την περιφερειακή ατζέντα και την ατζέντα των πόλεων, των αστικών κέντρων. Και μια ουσιαστική συμφωνία για την ανάπτυξη της περιφέρειας και της υπαίθρου θεωρούμε ότι είναι απολύτως σκόπιμη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα πλαίσια της Προεδρίας μας, στο πλαίσιο αυτό, θα αναρωτηθούμε σχετικά με την δημοσιονομική πτυχή της διαδικασίας αυτής. Θα οργανωθεί και σεμινάριο σε επίπεδο γενικών διευθυντών και διευθυντριών που προβλέπεται για τις 13 ενδεκάτου στην Βιέννη. Η διάδραση με την περιφερειακή και την αστική πτυχή τη πολιτική συνοχή θα αποτελέσουν επίση θέμα του σεμιναρίου. Αξιότιμε κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, στη διάρκεια τη Προεδρία μα θα πράξουμε πάντο δυνατόν για να επιτύχουμε τις συνθήκες πλαίσια για μια βιώσιμη και αηφόρο πολιτική συνοχής. Η συζήτηση για τις νομοθετικές προτάσεις θα διεξαχθεί σε όλα τα επίπεδα του Συμβουλίου πάντοτε σε στενή ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους φορείς. Το επόμενο εξάμεινο θα είμαστε η κινητήρια δύναμη για την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών στόχων. Εκτός από τον ρόλο μας συντονιστριών και συντονιστών, θα είμαστε ειλικρινείς οι διαμεσολαβητές και γεφυροποιοί. Έχουμε προετοιμαστεί καλά, έχουμε βάλει στόχους και έχουμε την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να τις επιτύχουμε σε κοινή προσπάθεια με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ως δείγμα ισχύω της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας βλέπω τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτου, το οποίο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει ότι μεταφέρει τη γνώμη και τις απόψεις των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Με την ομοσπονδική μας Υπουργό, κυρία Κέστιγκερ, η οποία επίσης υπήρξε Ευρωβουλευτής, θα, στο πρόσωπό της δηλαδή, θα βρείτε έναν συνομιλητή που γνωρίζει απολύτως την σημασία των γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ ως αντικαταστάτριά της θα προσπαθήσω στους επόμενους δύο μήνες, που θα διαρκέσει δηλαδή η άδεια μητρότητά της, ε, να ε, παίξω τον ρόλο αυτό. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και είμαι στην διάθεσή σα για ερωτήσει και απαντήσει. Απαντήσει που θα προσπαθήσω να δώσω με πλήρη συνείδηση του τι θα έλεγε η Υπουργός μας κυρία Κέστιγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις μας. Ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τους συντονιστές. Ο κύριος Μπάντης, Thank you. Thank you very much. Ο κύριος Βανίστελρο, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τα καλά νέα. Ε, για το γιο, πώς λέγεται. Johannes δύο ονόματα, ωραίο χριστιανικό υπόβαθρο μάλλον. Ε, ε μεταφέρετε έτσι τις καλύτερες ευχές μας όλων μας ε, εδώ από απόσταση θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι ελπίζω όλα να πάνε κατευχήν τώρα για την ε, προεδρία σας αναλαμβάνετε από τη Βουλγαρική Προεδρία έχουν γίνει ήδη πολλά Έχουμε φτάσει σε κανονική ταχύτητα πορείας. Έχετε τους γενικούς κανονισμούς που αναφέρατε και σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έχετε αναφέρει δύο πράγματα στο πρόγραμμα εργασιών σας. Λέτε ότι θα επιταχύνετε. Λέτε ότι θα επιδιώξετε γρήγορη ε, πρόοδο όσον αφορά το διαπραγματευτικό πακέτο και λέτε ότι Πιθανότατα θα λάβει χώρα μια συνάντηση τον Νοέμβριο. Και κοιτώντα αυτά τα 40, τις 40 σελίδες δραστηριοτήτων, δεν βρήκα πολλά πράγματα για τη συνοχή. Για να είμαι ειλικρινής, μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Είναι άτυπη υπουργική για τη συνοχή ή ευρύτερη. Γιατί είδα ότι gag meeting η αποσίδα, γιατί σε τέτοιου είδου δραστηριότητε κάθε προεδρία ε, μα λέει ότι ναι, έχουμε συμφωνία για το πού βρισκόμαστε, πού θα κληθούμε. Να ανταλλάξουμε απόψει. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά από την πολύ επιτυχή διήμερη στη Σόφια που είχαμε για την πολιτική αυτή. Θα μπορούσατε λοιπόν να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Έχω βρει τώρα μια ημερομηνία 13 Νοεμβρίου. Ε, ποια ήταν η θέση του Κοινοβουλίου. Μιλάτε για ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Είμαστε το Κοινοβούλιο, ναι. Και μετά γενικά μπορείτε να μας πείτε κάτι δεν βρήκα κάτι για τη στρατηγική για τις Άλπεις. Για τις μακροπεριφέρειες. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε λίγο. Την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή εγώ βρέθηκα σε μια συνάντηση στο Ίνσπρουκ την εβδομάδα των καινοτόμων περιφερειών. Και εκεί είδα ότι ο τρόπος ε, που ακολουθεί η Αυστρία και οι άλλες περιφέρειες ε, που εκπροσωπούνταν εκεί για την ε, αποδοχή των κονδυλίων ε, αφορά ουσιαστικά τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ε, νέων τεχνολογιών, ε, νέας οικονομίας. Πήγα στο υπολογιστικό κέντρο στο Ινσμπρουκ. Εμβληματική, εμβληματικό έργο. Αλλά όπως είδαμε έχει ξοδέψει τόσα πολλά χρήματα από το Horizon 2020 η Ευρώπη. Αλλά οι εταιρείε δεν είναι μέλη αυτή αυτή τη μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, αν συγκρίνουμε με το Ισραήλ, την Κίνα και τι ΗΠΑ, δεν είμαστε παρά μια στάλα στον ωκεανό. Με λίγη περισσότερη λοιπόν συγκέντρωση μπορούμε να κάνουμε τα, παντού τα ίδια πράγματα. Αλλά στην περιφερειακή πολιτική έχετε και την προσέγγιση τη έξυπνη ε, ειδίκευση. Οπότε επιτρέψουμε στου πρωτοπόρου να του δώσουμε τη δυνατότητα να συνεργάζονται καλύτερα και σε όσου ακολουθούν να τους ε, πούμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται όχι μόνο ταχύτητα αλλά και ειδικότητε. Αν λοιπόν ε, το έχετε υιοθετήσει αυτό, πείτε μας πώς. Εξηγήστε μας τη φιλοσοφία σας. Αλλά κατά τα άλλα το πρόγραμμα εργασιών σας ε, δεν λέει πολλά για την πολιτική συνοχή. Μήπως υπάρχει κάποια έκπληξη, μας επιφυλάσσετε κάποια έκπληξη στις προσκλήσεις που έχετε απευθύνει προς το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Βαν συντονιστής του ΕΛΚ, η κυρία Κρέλ, συντονίστρια των Σοσιαλδημοκρατών. Κυρία Κρέλ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω σήμερα και βεβαίως δικαίως είπατε ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς ενδιαφέροντος και εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να επιταχύνει, να εργαστεί ως το δυνατόν ταχύτερα, χωρίς βέβαια να μειώσει την ποιότητα των συζητήσεων, αλλά στο προσωρινό μας χρονοδιάγραμμα έχουμε βασιστεί στην ιδέα ότι ίσως ήδη τέλη του έτους μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και έτοιμες και να διεξαχθούν ήδη μέσα στο έτος κάποιοι τριμμυρίσεις διάλογοι. Ποια είναι η εκτίμησή σας, είναι η Προεδρία σε κατάσταση να ξεκινήσει κάτι τι τέτοιο τον Δεκέμβριο. Έχετε σχετική εντολή ή απλώς συζητούμε. Διότι εάν είναι έτσι, αν δηλαδή απλώς συζητήσεις κάνουμε, δεν χρειάζεται ε, να βιαστούμε. Μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτούς περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να μάθουμε αν η Προεδρία είναι όντως προετοιμασμένη και μπορεί να μπει σε πραγματικούς γνήσιους τριμερείς διαλόγους. Επιτρέψτε μου και μια ερώτηση. Αναφερθήκατε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σωστά. Δεν μπορούμε να δώσουμε τελική μορφή ακόμα σε κανονισμούς σχετικούς, αλλά θυμούμε ότι η Αυστρία δήλωσε σαφώς ότι η Αυστρία επιθυμεί να λάβει πολλά χρήματα, δεν θέλει όμως να πληρώσει πια πολλά χρήματα. Και δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με τις προτάσεις Oettinger για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, προτάσεις τη Κομισιόν δηλαδή. Πολύ λιγότερο δε να ακολουθήσει τι φιλόδοξε προθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να μα πείτε κάτι σχετικό, διότι αυτό βεβαίω έχει σημαντικέ επιπτώσει στην πολιτική συνοχή. Λέτε ότι είναι περίπου το 1 τρίτο του συνολικού προπολογισμού, αλλά στην πολιτική συνοχή αναμένουμε περικοπέ τη τάξη του 10%. Και τι θα πει αναμένουμε, είναι ήδη μέσα στην πρόταση τη επιτροπή. Και αυτό σημαίνει εν ώψη και των δυσχερών προκλήσεων και σε πολιτικές που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτική συνοχή όπως προστασία του κλίματος, όπως έρευνα, όπως καινοτομία, όπως ψηφιοποίηση που όλα αυτά όμως πρέπει να, να χρηματοδοτηθούν και από την πολιτική συνοχή. 10% περικοπές δεν είναι και λίγες. Μήπως μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτού. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ms. on behalf... Ευχαριστούμε η κυρία Τόμασιτς εκ μέρους του ECR. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, οι νέες χώρες μέλη παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά λιγότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί αρκετά. Μπορείτε να, μιλήσει, να πείτε μάλλον πως ε, θα γινόταν να εξαντλήσουν περισσότερο τα οικονομικά μέσα από τα ευρωπαϊκά ταμεία οι νέες χώρες. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους της Άλντερ, κύριο Σμίτεμπλεκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ την Υπουργό και σας ευχαριστώ και για την ευελιξία σας που αντικαθιστάτε τη συναδερφό σας. Και η ομάδα μου τη εύχεται ό,τι καλύτερο για το νεογέννητο αγοράκι της. Κοίταξα το πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας και η επικουρικότητα δέκα φορές εμφανίζεται, ενώ η συνοχή δεν εμφανίζεται καθόλου. Το είπε και ο συνάδελφος από το ΕΛΚ, ο κύριο Φανίστερόι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Η αρχή της επικουρικότητας είναι η ταυτότητα που θα χρησιμοποιήσετε και θα έχετε και μια ε, διάσκεψη ψηλού επίπεδου Έχει να κάνει και με τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Θέλουμε να απαντήσετε γιατί ωραία είναι η επικουρικότητα, αλλά πιστεύουμε ότι δεν είναι λύση στα ευρωπαϊκά προβλήματα το να χρησιμοποιούμε τη λέξη επικουρικότητα, κυρίως με τα προβλήματα που έχουμε σήμερα που χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή από ποτέ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου. Και η δεύτερη έχει να κάνει με τη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Υπάρχει στο εγγραφό σας ότι θέλετε μια διαδικασία πιο αποτελεσματική διαπραγματεύσεων ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προς τα τέλη της χρονιάς. Τι σημαίνει αυτό, τι, ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν για σας και για την Αυστρία. Ενώ υπάρχουν νομικά και διοικητικά προβλήματα στα διασυνοριακά ζητήματα. Και τι λέτε για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασχοληθεί με την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού όταν ε, υπάρχουν ανεπάρκειες ε, στο κράτος δικαίου σε διάφορες χώρες μέλη. Στο Συμβούλιο αυτό συζητιέται μια κρυφή συζήτηση και εσείς ως Αυστριακή Προεδρία θα μπορούσατε να βοηθήσετε πολύ, να κάνετε ένα βήμα δηλαδή προς τα πρός και όπως είπατε και ίδια στο εγγραφό σας να περάσετε στη Ρουμανική Προεδρία που είναι η επόμενη ένα πλήρες πακέτο και καλά επεξεργασμένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν γίνει αυτό. Ευχαριστούμε κύριο Παπαδημούλης, εκ μέρου της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, τις ευχές μου για το νεογέννητο και από τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά επιτρέψτε μου να μπω στην ουσία του θέματος διάβασα τις δεκάδες σελίδες με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Για τις πολιτικές συνοχής δεν βρήκα σχεδόν τίποτα. Την ίδια τη λέξη συνοχή, δεν θυμάμαι αν την είδα καθόλου, άκουσα τον καγκελάριο Κούρτ στην Ολομέλεια πριν λίγες ημέρες. Δεν είπε ούτε μια φορά τη λέξη συνοχή, ενώ είπε πάρα πολλές φορές τη λέξη επικουρικότητα page 14. Page 14. once. Ευχαριστώ κύριε Βανιστερόι. Όσα λέτε επιβεβαιώνουν αυτό που ακριβώς είπα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου που λέει ούτε ένα ευρώ περικοπή στις πολιτικές συνοχής. Πώς την βλέπει η Αυστριακή Προεδρία. Γιατί στα χρόνια που πέρασαν έχουν αυξηθεί επικίνδυνα οι ανισότητες μέσα στην Ευρώπη. Και οι κοινωνικές και οι περιφερειακές. Είσαστε υπέρ ή κατά τις θέσεις που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης μαθαίνω ότι η Αυστρία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντίθετη ακόμη και με την πρόταση της Κομισιόν που λέει 10% περικοπές για τις πολιτικές συνοχής. Θέλετε περισσότερες περικοπές και από την πρόταση Οέτιγκερ. Μας λέτε ότι θα οργανώσετε μια συνάντηση στο τέλος, στα μέσα του Νοεμβρίου. Με ποιες προτάσεις θα πάτε σε αυτή την στη συνάντηση ως Αυστριακή Προεδρία. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις σε αυτά, γιατί εδώ η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής στη συντριπτική της πλειοψηφία, κυρία Υπουργέ, ανεξαρτήτως πολιτικών οικογενειών, θέλει ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, υπερασπίζεται την πολιτική συνοχής και δεν θέλει την υπονόμευση και την αποδυνάμωση των πολιτικών συνοχής. Το ακούσατε και από τους συντονιστές του EPP, του ALDE, των σοσιαλιστών και θα ήθελα σε αυτά τα θέματα όσο δυνατόν σαφέστερες απαντήσεις γιατί η ασάφεια φαίνεται να θυμίζει ροκάνισμα χρόνου. Να περάσουμε το θέμα χωρίς να γίνει τίποτα στη Ρουμανική Προεδρία. Thank you, Miss Vanna. Ευχαριστούμε. Κύριε Βάνα, μέρος των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας απευθύνω το καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ ε, τώρα στην Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως, διότι είπαμε και το πρωί στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και βεβαίω ε, τι πλέον εγκάρδιες ευχέ μου στην Υπουργό σα, κυρία Κέστιγκερ. Δεν είναι και εύκολος ο τομέα που έχετε αναλάβει για του επόμενου δύο μήνες και γι' αυτό είστε σήμερα βεβαίως παρούσα εδώ. Η ε, περιφερειακή ανάπτυξη είναι από τα πιο περίπλοκα θέματα που θα συζητήσουμε του επόμενου μήνες και γι' αυτό συμφωνώ απολύτω με όσου μίλησαν προηγουμένω και είμαι και εγώ κατάπληκτη, διότι στο υποβληθέν πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας έξι γραμμές, έξι σειρές αναφέρεται μονάχα για την πολιτική της συνοχής. Δεν το είπατε σήμερα εδώ, βέβαια το σύνθημα της ε, Προεδρίας σας είναι η Ευρώπη που προστατεύει. Ωραίο σύνθημα είναι αυτό, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι αυτή η Ευρώπη που προστατεύει στην πολιτική της Αυστριακής Προεδρίας μάλλον περιορίζεται σε ένα σύνολο θεμάτων που είναι προστασία εξωτερικών συνόρων, μεταναστευτικό, άμυνα. Αυτό που βλέπουμε να λείπει είναι κάποιες προτεραιότητες της κοινωνικής προστασίας, της προστασίας των εργαζόμενων και της προστασίας του κλίματος που έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και στην πολιτική της συνοχής. Γι' αυτό η πρώτη μου ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δέσμευση 30% για στόχους προστασίας του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ένα στόχο 25%. Ποια είναι η θέση της Αυστριακής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδιακή Αυστριακή Κυβέρνηση, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Κρέρ άλλωστε, στο ζήτημα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα το πω διπλωματικά, είναι μάλλον υπέρ μιας περιοριστικής στάσης, το λέω προσεκτικά και πάλι που ε, για μας δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Η αυστριακή κυβέρνηση προσπαθεί ε, να προωθήσει την πρόταση του 1% που είναι ακόμα χαμηλότερη από τις προτάσεις του Επιτρόπου Έτιγκερ και είναι μάλλον λοιπόν, συμπαρατάστε μάλλον με τις χώρες που πλοκάρουν. Πώς θα καταρρίξουμε, από τη μια μεριά ζητούν λιγότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από την άλλη μεριά όμως προσπαθούν να διατηρήσουν τις ίδιες καταβολές κονδυλίων υπέρ των αγροτών στην Αυστρία. Αυτό εμένα μου μυρίζει λαϊκισμό. Είστε και υπουργό για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών. Και εγώ είμαι συντονίστρια στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Γι' αυτό έχω και ένα ερώτημα για αυτήν την υπόθεση. Μας ανησυχεί το ότι στο CPR η οριζόντια αρχή της ισότητας φύλων και της αποφυγής διακρίσεων κάπου φαίνεται να έχει χαθεί. Πώς θα φροντίσετε ώστε, το mainstreaming της ισότητας των φύλων να συνεχίσει να μπαίνει οριζόντια σε όλες τις πολιτικές. Και βεβαίως και η αποφυγή διακρίσεων. Και τι γίνεται και με το βάθεμα της αρχής της εταιρική σχέσης, της συνεργασίας με συμπερίληψη τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων, κοινωνικών εταίρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Συμμετοχή όλων αυτών στην αξιολόγηση των διαθροτικών ταμείων. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού και ποια βήματα πρόκειται να κάνετε για το βάθεμα της αρχής, της εφαρμογής δηλαδή, της αρχής της εταιρικής αυτής συνεργασίας. Σε αυτές τις έξι γραμμές στο πρόγραμμά σας που αναφέρετε ως προτεραιότητα, μιλείτε για την απλοποίηση. Απλοποίηση Βέβαια, η χ καλά και εμεί, οι πράσινοι είμαστε υπέρ τη απλοποίησης. Όμως υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνο απλοποίηση να συμπαρασύρει και κάποιες σημαντικές πολιτικές αρχές, όπως αυτές που είπα, gender mainstreaming και αποφυγή διακρίσεων. Από την άλλη μεριά, με το σύνθημα της επικουρικότητας που φέρνετε εσείς σαν δεύτερο στόχο σα και κάτω από το μανδύα αυτής της θετικής προσέγγισης περισσότερα δικαιώματα υπέρ πόλεων, δήμων, κοινοτήτων κλπ. Όμως, όποιος εξετάσει το πρόγραμμά σας θα δει ότι πίσω από το σύνθημα της επικουρικότητας κρύβεται κάποια επανεθνικοποίηση και στην πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και αλλού. Γι' αυτό σας ερωτώ, δεν βλέπετε καθόλου τον κίνδυνο αυτό. Και στην ενίσχυση της αρχής της επικουρικότητας δεν βλέπετε καμία επαναφορά αρμοδιοτήτων από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο περιφερειακό και κοινοτικό τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να απαντήσετε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Έχω δύο νόματα στις άλλες ερωτήσεις. Υπάρχει κανένας άλλος που θέλει το λόγο. Ωραία. Συνεχίζουμε με τους δύο. Ε, η κυρία Σμίτ πρώτα απ' όλα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Δεν είναι βέβαια εύκολο το έργο σας να είστε παρούσα εδώ και να αντικαθιστάτε την Ελισάβετ Κέστινγκερ σε ένα τόσο ευρύ και δύσκολο θέμα. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συνεργασία σας. Τα κονδύλια της συνοχή είναι αυτά που καταλήγουν πραγματικά στον πολίτη και το νιώθει ο πολίτης αυτό. Γι' αυτό και για μας έχουν μεγάλη σημασία. Γνωρίζουμε ποια είναι τα δύσκολα θέματα και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε και εσείς τους επόμενους μήνες. Πολιετές, δημοσιονομικό πλαίσιο. Γι' αυτό έχω δύο τεχνικού χαρακτήρα ερωτήματα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τώρα η το ποσοστό συγχρηματοδότησης υπολογιζόταν σύμφωνα με το κατακεφαλή ΑΕΠ. Τώρα υποτίθεται θα αλλάξει. Θα περιληφθούν παράγοντες όπως μεταναστευτικό, αλλαγή κλίματος κλπ. ως κριτήρια. Ερώτηση λοιπόν. Πώς βλέπετε αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρείτε ότι θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί πλειοψηφία υπέρ των ιδεών αυτών στο Συμβούλιο. Δεύτερο, τα κονδύλια συνοχή, πάλι σύμφωνα με την πρόταση τη Κομισιόν, θα συνδεθούν με κάποια αιρεσιμότητα. Την διατήρηση του κράτους δικαίου, όπου εδώ κάποια προβλήματα αναφύονται σε κάποιες χώρες μέλη και με ενδιαφέρει εδώ εάν ο μοχλό αυτός, κατά τη γνώμη σου, έχει πιθανότητα να ισχύσει, να εφαρμοστεί για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού που ταξιδεύει, μεταβαίνει σε αποστολές και εξετάζει επιτόπου έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από κονδύλια συνοχής. Έχω απολύτως δική μου άποψη σε ό,τι αφορά τις προτάσεις Oettinger. Θεωρώ ωστόσο ότι θα είναι δυνατό να γίνουν κάποιες εξοικονομήσεις εδώ και εκεί. Όμως, οφείλω να πω, για να επανέλθω σε αυτά που είπα στην αρχή, ότι απλοποίηση των προγραμμάτων στήριξης είναι απόλυτα σημαντική και, ξαναλέω, τα κονδύλια συνοχής είναι τα χρήματα εκείνα τα οποία βλέπει και νιώθει ο πολίτη οι διάφορε χώρε μέλη να φτάνουν μέχρι την καθημερινή του ζωή. Ευχαριστώ για τι απαντήσει που θα δώσει. Και εμεί ευχαριστούμε. Ο κύριο Μοσκούρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την ε, Υπουργό για τους προσανατολισμούς που μας ε, εξήγησε και που θα προθεθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Αυστιακής. Θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, ξέρουμε ότι είναι και το μεταναστευτικό που θα μας απασχολήσει, αλλά και το χάσμα το οποίο μεγαλώνει ανάμεσα στους καθαρούς συνεισφορείς και εκείνους που επωφελούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Είμαστε σε μια στιγμή αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον που θέλουμε να προσφέρουμε στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Το υπενθυμίσατε και εσείς στην παρέμβασή σας ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο μέσο επένδυσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και των περιφερειών. Βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Χωρίς αυτή την αλληλεγγύη, οι ανισότητες μεταξύ περιφερειών θα ενισχυθούν και οι συμπολίτες μας από τις λιγότερο ευνοημένες ε, περιφέρειες θα βρεθούν σε δινή θέση όπως ε, εκείνοι που ζουν στις άκρος περιφερειακές περιοχές. Γι' αυτό και το ακούσαμε και πριν, υπάρχει ο φόβος της μείωσης των κονδυλίων που οδηγεί σε απογοήτευση αφενός, αλλά από την άλλη δύσκολα μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί μόνο η πολιτική συνοχής προσφέρει απτά αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική συνοχής λοιπόν να αποτελεί μια μεταβλητή η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Βασιζόμαστε λοιπόν σε εσά και στις δικές σας αρμοδιότητες για να προχωρήσετε σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε σε φιλόδοξα αποτελέσματα. Να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε να βασίζεστε στη δικιά μας επικοδομητική συνεργασία, αλλά και στην αποφασιστικότητά μας επίσης, προκειμένου να προχωρήσουμε με μια πολιτική συνοχής ισχυρή και στο ύψος των ε, προκλήσεων που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις και τα σχόλια των μελών της Επιτροπής ε, Ρέγγι και των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Σας δίνω τώρα το λόγο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω χωρίζοντας τις σε ομάδες, γιατί ορισμένες ερωτήσεις επαναλήφθηκαν. Όσον αφορά την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην συνάντηση του Νοεμβρίου το οποίο θα διεξαχθεί, η οποία μάλλον θα διεξαχθεί σε επίπεδο Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Πρόκειται για συνάντηση που θα γίνει σε επίπεδο Υπουργών Συνοχής. Για την ώρα δεν έχουν προβλεφθεί άλλες συνεδριάσεις. Βεβαίως θα υπάρχει πληροφόρηση Γνωρίζετε ότι μπαίνουμε σε νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει για το 2021 έως 2027 και κάθε θεσμικό όργανο έχει τους σχετικούς κανόνες που διέπουν τις εργασίες του. Η άλλη ερώτηση αναφερόταν στους τριμερείς διαλόγους. Δεν θα είναι δυνατόν να έχουμε εντολή για όλους τους τριμερείς διαλόγους αλλά θα είναι δυνατόν να δοθεί μερική εντολή για ορισμένους. Α, ποια ήταν η άλλη σας ερώτηση. Ποια μέρη θα έχουν εντολή, ρωτάει η κυρία Κρέλ. Αυτό θα το δούμε και θα σας ενημερώσουμε. Μετά ήταν η ερώτηση Ευρώπη που προστατεύει. Η Ευρώπη που προστατεύει, για μένα αυτό σημαίνει και το δηλώνω ρητά, ότι δεν πρόκειται μονάχα για προστασία κατά της ε, παράτυπης μετανάστευσης. Σύνθημα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας σημαίνει αντιμετώπιση όλων των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και εδώ συγκαταλέγω προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση, οι συνέπειες πολεμικών σειράξεων στη γειτονιά μας, αλλά και η εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού και όπως λέχθηκε άλλωστε σήμερα και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και αυτά μας απασχολούν. Και ιδίως ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων του μεταναστευτικού, της ενσωμάτωσης, της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βεβαίως και στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Ορισμένοι ημών θίξατε και μου ζητήσατε να σχολιάσω την αυστριακή οπτική επί των θεμάτων αυτών. Εγώ βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα ως Προεδρεύουν του Συμβουλίου, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Άρα δεν θα μιλήσω για εθνικά θέματα. Θα μιλήσω μόνο για τα θέματα που απασχολούν το Συμβούλιο. Επίσης το θέμα της χρηματοδότησης τέθηκε από εσά ορισμένες φορές. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συζητείται και διαπραγματεύεται επ' αυτού ο συνάδελφός μου Μπλούμε στο επίπεδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών και ιδίω ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της ανατομέα νομοθεσίας. Όπως είπα, ο συνάδελφός μου Μπλούμε προεδρεύει του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων όπου συζητείται το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο συναντάτε και με προσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σύμφωνα με τα Ιωθώτα, ο πρόεδρός σας Ταγιάννη έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί ευθέως άμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Μετά με ρωτήσατε για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον χώρο των Άλπαιων και σχετικά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, που είναι ένα καινοτόμο μοντέλο της περιφερειακής συνεργασίας για επιλεγμένα θέματα αναπτύξεως, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Αυστρία για τον χώρο των Άλπαιων και του Δουνάβεως η υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών, ιδίω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή Περιφερειών, θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μα και θα πρέπει να συνεχιστεί. Άκουσα μετά την ερώτηση σχετικά με το πού θα στραφεί, που θα πρέπει να στραφεί η στόχευση της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι μπορώ να δώσω την καθαρή απάντηση ότι η στόχευση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι οι πιο φτωχές περιφέρειες και κράτη. Για τον μηχανισμό των διαμεθοριακών επιλύσεων διαφορών. Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασφαλώς είναι αναγκαία για τις παραμεθόριες περιοχές. Για την ώρα πάντως είναι αρκετά περίπλοκη η προτινόμενη αυτή ρύθμιση. Ευχαρίστως να προχωρήσουμε σε κοινή συζήτηση με τους εισηγητές σας και η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί με συμμετοχή μελών της ομάδας μας τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Α, ναι, ναι, μένει ακόμα το ζήτημα της ισότητας των φύλων gender mainstream. Βεβαίως, θα ήθελα να πω εδώ ότι οι οριζόντιοι στόχοι με κανένα τρόπο δεν έχουν χαθεί. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιλεξιμότητος έργων, δεν έχουν χαθεί. Το ίδιο και η αρχή της εταιρική συνεργασίας. Και ο κώδικας διοντολογίας της περίοδου 2014 2014-2020 παραμένει και θα παραμείνει και για το μέλλον ισχυρός. Και θα ήθελα βέβαια επειδή θίξατε το θέμα και επειδή το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ιδίω η δικαιοσύνη απέναντι στα δύο φύλλα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας και αποτελεί και πρέπει να ξαναγίνει προτεραιότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ώρα δεν υπάρχει καμιά σχετική στρατηγική. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα στρατηγική για την δικαιοσύνη απέναντι των φίλων. Μιλήσατε και για την επικουρικότητα. Η Ευρώπη και εμείς είμαστε Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη λοιπόν υπάρχει για να λύνει τα μεγάλα προβλήματα, ώστε οι πολίτες αμφωτέρων των φύλων να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στην Ευρώπη, να αισθάνονται ασφαλείς ως Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες. Όμως ορισμένα πράγματα μπορούν να λυθούν καλύτερα επί τόπου. Και γι' αυτό εμείς λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη την επικουρικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Θα δώσω το λόγο στους συναδέρφους για κάποια σχόλια και παρατηρήσεις. Γιατί για μας στην Επιτροπή Ρέγγι η σημερινή συζήτηση έχει τεράστια σημασία. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε τις εργασίες μας, να τις οργανώσουμε μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογέ. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα επικεντρωμένοι σε αυτά τα ζητήματα και προσπαθούμε να κάνουμε θαύματα, όπως είπε ένας συνάδελφος λίγο νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό, συνεπώ, να ξέρουμε ποια είναι η θέση τη Αυστριακή Προεδρία. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρέλ και μετά στον κύριο Φανίστερόι. Κυρία Κρέλ. Η κυρία Κρέλ, μία παρατήρηση και μία ερώτηση ακόμη. Η παρατήρηση είναι η εξή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που μιλούμε στα πλαίσια της συνομοθετικής διαδικασίας που μιλούμε για συνοχή λοιπόν, όπου μια Προεδρία δεν μας προσκαλεί, δεν προσκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση. Ε, αισθάνομαι κάπως παράξενα. Ίσως όμως να υπάρχει και κάποια παρανόηση. Η ερώτησή μου, και επανέρχομαι στην αρχική μου ερώτηση με άλλη διατύπωση, η Αυστριακή Προεδρία βλέπει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και να συμβάλλει σε μια το δυνατόν ταχύτερη λύση στα πλαίσια του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε κύριο Φανίστεροι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αλλά λίγο πολύ και εγώ αυτά σκέφτομαι που είπε και η κυρία Κρέλ. Δηλαδή κάθε ανταλλαγή στο παρελθόν, αλλά ίσως να υπάρχει αλλαγή, είναι μια πρόσκληση για συμμετοχή. Εγώ πήγα για δικό μου λογαριασμό, αλλά εσείς είπατε ότι πρόκειται για συνάντηση υπουργών. Ναι, αλλά πώς το οργανώνετε αυτό. Δεν είσαστε μόνο προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Πώς ε, οργανώνετε αυτή την επαφή, την επικοινωνία θυμάμαι, εντάξει, ούτε η Ολλανδία ούτε κι εσείς είστε χώρες συνοχής, αλλά θυμάμαι ότι στο Άμστερνταμ φροντίσαμε να δουλέψουμε για τις πόλεις. Δραστηριοποιηθήκαμε πολύ, ενώ από αυτά που μας λέτε εσείς, δεν βλέπουμε ότι θέλετε να δουλέψετε πάνω σε αυτό. Οπότε δεν βλέπω από πού θα έρθει έμπνευση. Πού είναι η πρόσκληση. Δεν τη βλέπω. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία προεδρία να αρνείται το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έναν τρόπο που εγώ τον εκλαμβάνω περίπου ως προσβλητικό και η οποία να αποφεύγει να ανοίξει και τα χαρτιά της για το πώς βλέπει αυτά τα θέματα που μας απασχολούν σας ρωτήσαμε πώς βλέπετε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές συνοχής στο πλαίσιο του νέου MFF, του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν μας είπατε τίποτα. Μας παραπέψατε σε ένα συνάδελφό σας, ο οποίος όμως δεν είναι εδώ. Σας ρωτήσαμε πώς βλέπετε τις προτάσεις Σέτιγκερ, που έχουν περικοπές 10% για τα κονδύλια συνοχής, μας παραπέψατε πάλι στον ίδιο απόντα συνάδελφό σας. Εμείς όμως έχουμε εσάς εδώ, θα μας πείτε πώς βλέπετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις θέσεις του, αντί να μας αποκλείεται από τις μελλοντικέ συναντήσεις. Δεν μου έχει ξανατύχει τέτοια προεδρία τόσο εχθρική και προσβλητική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε τις παρατηρήσεις, δεχτείτε σαν έτσι φορτισμένες, επειδή ακριβώς μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η περιφερειακή πολιτική για το μέλλον. Όλοι οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, εμπλέκονται πάρα πολύ και γι' αυτό βλέπετε αυτή τη συναισθηματική φόρτιση. Περιμένουμε πώς και πώς τέτοιες ανταλλαγές απόψεων μαζί σας. Οπότε να μεταφέρετε και στο συνάδελφό σας τα σχόλια και εντάξει, απαντήστε παρακαλώ σε ό,τι σχόλια μπορείτε. Υπουργό. Κατανοώ ότι επανέρχεστε σε κάποια ερωτήματα. Νομίζω όμως ότι όπως είπα και προηγουμένως, το πολιτεύστημο δημοσιονομικό πλαίσιο εξακολουθεί να ευρίσκεται υποσυζήτηση. Εγώ βρίσκομαι εδώ ως Προεδρία και για το λόγο αυτό δεν επιθυμώ να συζητήσω εθνικά θέματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να δούμε βέβαια το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων, να γνωρίζουμε εν τέλει πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για την πολιτική της συνοχής, ώστε όντως να μπορέσουν να διατεθούν τα κονδύλια αυτά για την πολιτική συνοχής. Να επανέλθω στο δικό σας ερώτημα, κυρία Κρέλ, σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Νοεμβρίου, θα είναι συμβούλιο γενικών υποθέσεων. Δηλαδή πρόκειται για επίσημο συμβούλιο, όχι ανεπίσημο. Στο επίσημο συμβούλιο προβλέπεται ότι συμμετέχουν υπουργοί. Και επομένως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στις επίσημες αυτές διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς και τις υπουργούς συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η ενταλλαγή απόψεων με την εκπρόσωπο της Αυστριακής Προεδρίας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους για κάποια από τα θέματα ενδεχομένως, ίσως και όχι. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή μας. Θερμούς χαιρετισμού στους συναδέλφους σας και συγχαρητήρια για το νεογέννητο μωρό και ελπίζω να είναι επικοδομητική η Αυστριακή Προεδρία. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Στις 29 Μαΐου φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρότασή της για ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Μπορώ να παρακαλέσω <laughs> Uh, λοιπόν, ξαναπροσπαθώ για να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Συνεχίζουμε τώρα τη συζήτησή μας και θα κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε ουσιαστικά επί της γνωμοδότησής μας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΠΛΑΣ. Στι 29 Μαΐου Φέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε την πρόταση για το νέο Ευρω... Ε, κοινωνικό Ταμείο ε, Plus. Στις 11 Ιουνίου ο Πρόεδρος παρέπεψε την πρόταση αυτή στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Ρέτζη είναι μία από τις επιτροπές που είναι αρμόδια για τη σύνταξη γνωμοδότησης. Η κυρία Μπρέσο έχει συντάξει μια πρώτη άποψη για αυτή την ε, γνωμοδότηση για τη σημερινές συνεδρία και θα ανταλλάξουμε σήμερα απόψεις. Η συγκίτρια προτείνει να παρουσιάσει το σχέδιο χρωμοδότησής της στις 3 Σεπτεμβρίου, σωστά. Πολύ ωραία και θα την ψηφίσουμε σε μια από τις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Πιθανότητα τον Οκτώβριο. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα υιοθετήσει την, τελευταία της, την τελική της έκθεση της 27 Νοεμβρίου. Δίνω το λόγο στην κυρία Μπρέσο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως υπενθυμίσατε κι εσείς, αυτό ισχύει κάπως για όλες τις εκθέσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα περιορισμένου χρόνου. Όλοι οι εισηγητές, οι κύριοι εισηγητές, ε, έχουν πίεση για να προχωρήσουν ε, στα γρήγορα. Εμείς φυσικά δεσμευόμαστε από τους χρόνους της ε, Επιτροπής ΕΜΠΛΕ. Εγώ έχω ήδη επισημάνει στην εισηγήτρια της Επιτροπής ότι σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει κάποιο συντονισμός μεταξύ του γενικού κανονισμού, του κανονισμού ε, κοινών διατάξεων και των κανονισμών που αφορούν τα επιμέρους εμείς δηλαδή ξεκινάμε να, τις εργασίες μας, αλλά έχουμε πολύ στενά περιθώρια νομίζουμε. Δεν φαίνεται εύκολο να μπορούμε πρώτα να υιοθετήσουμε τους κανονισμούς για τα επιμέρους ταμεία και στη συνέχεια τον γενικό κανονισμό. Το λέω εδώ για να το ακούσουν και οι συγητές μας. Ε, πιο συγκεκριμένα για τον κανονισμό κοινών διατάξεων. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γνωρίζετε ότι είναι το κύριο μέσο της Ένωσης προς υποστήριξη της απασχόλησης, προς αρρωγή προς ε, ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας για την επένδυση συνολικά στο Ευρωπαϊκό Ανθρώπινο Κεφάλαιο. Η πρόταση που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή προβλέπει ότι πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα συγχωνευτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Πλάσα η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Στήριξης ε, για τους άπορους και το πρόγραμμα της κοινωνικής κοινοτομίας και το πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας. Το πλάς δηλαδή σημαίνει πολλά ταμεία συγχωνευμένα μαζί σε ε, έναν ενιαίο κανονισμό. Προφανώς, όπως υπενθύμισα με τη σειρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus αποτελεί κομμάτι μια σειράς διαρθρωτικών ταμεία που στο σύνολό του συνθέτουν τα ευρωπαϊκά επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία και αποτελούν κομμάτι του ε, κανονισμού κοινών διατάξεων. Δηλαδή βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια σειρά από σαν ε, μπάμπουσκες που περιλαμβάνουν η μία την άλλη. Γι' αυτό το λόγο οι χρόνοι ε, υιοθέτηση θα πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Εγώ θα υποστηρίξω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συνεχίσει να επιτελεί λωρό κλειδί στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας και στην πρόθεση της κοινωνικής ένταξης. Ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες, τους νέους, τους μακροχρόνια ανέργους, τους ανθρώπους με αναπηρία με αυτούς δηλαδή ως επίκεντρο. Προφανώς ε, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της ανάπτυξης δεξιοτήτων ε, και η έξυπνη εξειδίκευση ένας από τους βασικούς μας στόχους. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται και το άλλο θέμα που αποτελεί μία από τις στρατηγικές ε, κατευθύνσεις που έχει υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η περιβαλλοντική αηφορία, η κλιματική αλλαγή. Η έξυπνη λοιπόν εξειδίκευση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και όλες οι σχετικές ε, πολιτικές ε, περιβαλλοντικής ε, βιωσιμότητας είναι οι δύο μεγάλες κατευθύνσεις όπου προφανώς το πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου που πρέπει να δημιουργήσει μοντέλα ε, κατάρτισης ε, θα πρέπει να αφορά αυτούς τους τομείς, αυτούς τους τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν επενδύσεις κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Φυσικά, σημαντικό θα είναι η κατάρτιση να αφορά συγκεκριμένα ειδικότερα τους νέους χαμηλής κατάρτισης και που δεν βρίσκονται σε κάποιο πρόγραμμα ε, εκπαίδευσης ε, ή δεν εργάζονται, αλλά αφορά και διδάσκοντες, επιχειρηματίες, ερευνητές, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε, να στραφούμε προς τις κοινέ ε, προς τους κοινούς στόχους αυτούς θα πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η αλυσίδα ενδιαφερομένων. Κάτι που πρέπει να υπογραμμίσουμε, το οποίο δεν εμφανίζεται παρκώ στον κανονισμό όπως έχει σήμερα, είναι ότι πρέπει να δοθεί ένα σαφή ρόλος στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες ε, είναι αρχές δικαιούχοι αλλά και διαχειριστικέ. Συνεπώς πρέπει να αναφέρεται σαφώς στο νομοθετικό κείμενο αυτός ο ρόλος τους, ώστε να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι στα διαρθρωτικά ταμεία στο Ταμείο για την Περιφερειακή Πολιτική, στο Κοινωνικό Ταμείο. Ε, ουσιαστικά εκεί έχουμε δύο σκέλη μια αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρί ε, την προσαρμογή του ανθρώπινου κεφαλαίου στι ε, αναπτυξιακέ στρατηγικέ τη Ένωση, είναι σαν να μα λείπει το ένα σκέλο των διαρθρωτικών πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, προφανώ πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι πράγματι βλέπουμε θετικά την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου και για να γίνουν προσπάθειες ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του κοινωνικού ταμείου. Όπως πιθανότητα θα γνωρίζετε, αυτό ισχύει για όλα τα ταμεία, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη συνδέει ακόμα πιο άμεσα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις επενδύσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλαπλούς προγραμματικούς στόχους. Από τη μια πλευρά έχουμε κάποιους στόχους που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς ως πλαίσιο αναφοράς. Γενικό πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τις συστάσεις αναχώρα, τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν το πλαίσιο, συνθέτουν το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται τα διάφορα ταμεία και που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την, ε, ε, τη χάραξη των ε, προγραμμάτων. Από την άλλη υπάρχουν δύο κύρια προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Αφενός, οι προτεραιότητες που αναφέρονται για ολόκληρο το κομμάτι των διαρθρωτικών ταμείων, οι δύο προτεραιότητες που ανέφερα και οι άλλες πιο ειδικέ ε, του Κοινωνικού Ταμείου. Αφετέρου, σε αυτές προστίθεται στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κοινωνικού Ταμείου η αναφορά στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που ουσιαστικά ε, αντιπροσωπεύει σημαντικά όλες ε, οτιδήποτε αναφέρεται στα προγράμματα του Ταμείου μας. Το, τα εθνικά ε, επιχειρησιακά σχέδια και τα περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια εννοείται ότι πρέπει να παραμένουν εντός αυτού του πλαισίου στο οποίο αναφέρονται αυτά ε, τα διάφορα προγράμματα. Σε ένα προγραμματισμό που προφανώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πάντα αλλά και που πιο συγκεκριμένα πρέπει να αντιπροσωπεύει σε επίπεδο περιφερειών το συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο για τις περιφέρειες. Να υπενθυμίσω και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά έχουμε ένα 25% υψηλό ποσοστό δηλαδή του Ταμείου το οποίο θα πρέπει να δεσμευτεί για την κοινωνική ένταξη. Αφενός δηλαδή έχουμε τις παραδοσιακές πολιτικές κατάρτισης και εργασίας και αφετέρου έχουμε το θέμα της κοινωνικής ένταξης που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το ποσοστό αναφοράς στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων στις πιο συγκεκριμένες θεματολογίες της κοινωνικής ένταξης και σε αυτό προστίθεται ένα ποσοστό 2 έως 4%, 2% ελάχιστο 4% μέγιστο για τα άτομα σε που πάσχουν από υπερβολική ένδυα. Ε, περίπου το 30% των ε, συνολικών πόρων του Ταμείου θα δεσμευτούν για πολιτικές που σίγουρα είναι πολύ σημαντικές, αλλά και που δεν αποτελούν κομμάτι των παραδοσιακών κατευθύνσεων του κοινωνικού ταμείου. Και εκεί θα πρέπει να γίνουν εντατικέ προσπάθειες ε, με στόχο την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, ώστε να αποφευχθεί οι παραδοσιακές πολιτικές ε, εργασίας ε, να χάσουν σημασία. Αυτές είναι οι πρώτες μου παρατηρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρώτον θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά αυτούς τους νέους στόχους που προκύπτουν από τις διαπιστώσεις που έχουμε κάνει και παλιότερα ε, και σε όλες τις συζητήσεις ουσιαστικά αυτή την εποχή στη διαπίστωση ότι βρισκόμαστε ε, μπροστά σε μια κατάσταση ιδιαίτερης δυσκολίας ε, διότι σημαντικά ποσοστά του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρουν οπότε βοήθεια προς τους πλέον απόρους και γενικότερη βοήθεια για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να αυξηθεί. Αφετέρου, πρόκειται για μια πρόκληση που έρχεται να συμπληρώσει τις παραδοσιακές προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει το Κοινωνικό Ταμείο που όπως σημειώνεται ανέκαθεν προσανατολίζονταν στην κατάρτιση των εργαζομένων στις ενεργές πολιτικές εργασίες. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόκληση σημαντική. Και από αυτή την άψη λοιπόν το θέμα το ανησυχητικό των χρονοδιαγραμμάτων και του σωστού συντονισμού με τα άλλα ταμεία, τα διάφορα εργαλεία και τις ρυθμίσεις για τα άλλα ταμεία. Ε, αυτό το θέμα του συντονισμού λοιπόν με όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχαστεί. Έχουμε και την πρόκληση να συνεργαστούμε όλοι εντατικά, διότι όλο και περισσότερο όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία έχουμε και πλέον ε, να χαρακτηρίζονται και από γενικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο τους κλασικούς ε, που είχαμε συνηθίσει να λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό αποτελεί για μας αλλά κυρίως για τις ε, εκτελεστικές και διαχειριστικές αρχές μια πρόκληση που είναι αρκετά τρομακτική θα έλεγα δύσκολη και οι κύριοι συγητές μας το έχουν ε, υπενθυμίσει. Καλό θα ήταν πριν κλείσουμε να δούμε και τι γίνεται από άψη πόρων. Διότι η διαπραγματεύση για του συνολικού πόρου του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου είναι επίση πολύ σημαντική. Για να δούμε στη συνέχεια πώ πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο κάθε επιμέρου ταμείου θα μπορέσουν να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένε πολιτικέ. Διότι πάντα Μα ζητούν όλο και περισσότερο να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που έχει μπροστά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπρέσο για όλα όσα είπατε. Συγγνώμη για τους χρόνους, για το χρονοδιάγραμμα, όπως είπατε και εσείς. Εγώ λογικά θα μπορέσω να στείλω πριν από τις διακοπές ένα σχέδιο κειμένου στους συναδέλφους με μια πρώτη πρόταση τροπολογιών ε, για το κείμενο του κανονισμού ώστε όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές ε, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το κείμενο στην Επιτροπή και να ορίσουμε τους χρόνους για τις τροπολογίες. Οι συνάδελφοι πιστεύω ότι θα λάβουν εφόσον τα γραφεία της Κομισιόν μπορούν. Θα λάβουν το κείμενο λοιπόν πριν τις διακοπές έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε να μπορούν να ε, έχουν προλάβει να το δουν ε, έτσι μια δουλειά για τις διακοπές Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρέσο σαφέστατη η παρουσίασή σας για το θέμα και είμαστε νομίζω έτοιμοι έτσι με την γνωμοδότησή σας αυτή. Θα ακούσουμε τους ε, συντονιστές Έχουμε ήδη μια σαφή εικόνα για το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή μας. Το συστήσαμε και με τους συντονιστές ο κύριος Χέτμαν τώρα από τους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας αυτή. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται για απασχόληση και μάλιστα ποιότητα. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής και συμβάλλει και στην αηφόρο ανάπτυξη και στην πλήρη αξιοποίηση των πόρων των περιφερειών της Ένωσης. Η νομοθετική πρόταση για το πρόγραμμα αυτό προβλέπει και την ενσωμάτωση κονδυλίων προγραμμάτων τα οποία ως τώρα ήταν χωριστά. Το πρώην Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διάφορα προγράμματα υπέρ των νέων, προγράμματα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας και υγείας. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Σημαντικό πάντως είναι η συγκέντρωση αυτή των μέσων να ακολουθηθεί και από μια απλοποίηση. Πρέπει κανείς να τα αυτά προσεκτικά, αν δηλαδή είναι πράγματι οι βέλτιστες δυνατές προοπτικές και αν είναι και επαρκής. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να φτιάξει ένα νέο σχέδιο, το οποίο βεβαίως οδηγεί και σε διαφάνεια. Από την άποψη της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεως, βλέπω υπάρχουν μάλλον και δύο ε, συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού 100 για, τα περιφερε... για τις περιφερειακές περιοχές και 200 εκατομμύρια για προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης. Είναι σαφές ότι η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως σκοπό να συνδεθούν καλύτερα τα προγράμματα αυτά μέσω και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με τις συστάσεις αναχώρα αλλά και με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Αυτό θα βοηθήσει και, στην, και στις συστάσεις αναχώρα. Δεν είναι σαφές πόσα θα είναι τα κονδύλια. Κατά τη γνώμη μου θα είναι σκόπιμο να μελετήσουν το θέμα αυτό και να κάνουν μια ε, συγκεκριμένη ένα συγκεκριμένο υπολογισμό των κονδυλίων. Ελπίζω ότι σε συνεργασία με την εισηγήτρια θα μπορέσουμε να συντάξουμε το σχετικό έγγραφο το οποίο θα βοηθήσει και θα, αποτελέσει, θα συναποτελέσει βάση και τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Από το ΙΣΕΡ δεν έχουμε κανέναν. Άλντε τώρα, κύριος Μιλμπελ. Ευχαριστώ πολύ. Με ικανοποιεί η πρόταση τη Επιτροπή ουσιαστικά, γιατί νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία να μην ξεχνάμε στην Επιτροπή μα ότι δεν πρόκειται μόνο για επενδύσει, στην έρευνα, ε, αναπαλαίωση, πολιτιστική κληρονομιά κτλ. Αλλά πρόκειται επίση και πολύ σημαντικό επίση είναι να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό στην Ευρώπη. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύει πιστεύω ότι είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση του Κοινωνικού Ταμείου. Πρώτα απ' όλα συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό, όπως έχουν πει όλες οι πολιτικές ομάδες. Και το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω, αν βελτιώσουμε τις ε, οικονομίες επιδέσεων, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με λιγότερα χρήματα και καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας είναι κάτι πολύ σημαντικό για να καταρτιστεί κατάλληλα ο κόσμος και να μπορέσει έτσι να βρει τελικά δουλειά. Επίσης, με ικανοποιεί η συγχώνευση πέντε προγραμμάτων που σήμερα τα έχουμε ξεχωριστά το καθένα. Νομίζω ότι η προσέγγιση με το κοινωνικό ταμείο ΣΥΝ, το ESF+, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη και λυπάμαι γι' αυτό στη διαδικασία mainstreaming όσον αφορά το Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Εμείς θα θέλαμε και αυτό το ταμείο να συγχωνευτεί με το ESF+. Είναι μια χαμένη ευκαιρία αυτή, ενώ μιλάμε για αποτελεσματικότητα και απλοποίηση. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η συγχώνευση όλων αυτών των προγραμμάτων ελπίζω να μην είναι μόνο κάτι το διακοσμητικό, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαφορετικά κεφάλαια, διαφορετικά θέματα και να υπάρξουν συνέργειες και με άλλα προγράμματα. Το Horizon, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. Και τέλος, ο προπολογισμό για την διάσταση της υγείας, κατά τη γνώμη μου, είναι χαμηλότερο από ό,τι το σημερινό. Και με εκπλήσει αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για διασυνοριακή συνεργασία και στον τομέα της υγείας, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην υγεία, θα περίμενε κανείς μεγαλύτερο προϋπολογισμό για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας που θα βοηθήσει τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν ότι ο κόσμος εκπαιδεύεται καλύτερα για να μπορεί και να δουλεύει κάτω από καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Βάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά, κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την ε, συναδελφό μου Ράιντκε, η οποία είναι σκιώδη συγγήτρια. Το ESF sin ε, είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την επιτευξή του κοινωνικού πυλώνα. Στην ε, συγχώνευση σε ESF sin που αφορά διάφορα ταμεία όπως την πρωτοβουλία ε, για την νεότητα, το κοινωνικό ταμείο καθώς και άλλα, κοινωνική καινοτομία κλπ. Και βέβαια και τα προγράμματα υγείας. Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί προσοχή ώστε αυτό να μην επιβαρύνει τα μικρότερα προγράμματα με αποδυνάμωσή τους. Παραμένουν τα κοινωνικά μέτρα και ανέρχονται στα 25%. Εμείς οι πράσινοι είχαμε αγωνιστεί για το θέμα αυτό στην προηγούμενη ε, θητεία. Σημαντικό είναι επίσης τα 10% των κονδυλίων για την υποστήριξη νέων στις χώρες μέλη και ο στόχος που επιβάλλει στις χώρες μέλη για ένα ποσοστό του ESF υπέρ των πιο ευάλωτων ομάδων προσώπων μας φαίνεται πολύ θετικό. Τώρα, η κριτική που ασκούμε και θα σας ευνηδιάσει είναι η πολύ στενή διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Εκεί δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνες για τις οριζόντιες αρχές της ισότητας ανδρών και γυναικών και μη διακρίσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 της προτάσεως και στο Γενικό Κανονισμό ESF-SYN, αυτό μας φαίνεται θετικό. Και όπως και στη CPA e θα φροντίσουμε ώστε να μην προκύψει αποδυνάμωση αυτής της οριζόντιας αρχής της επόμενες διαπραγματεύσεις. Το ίδιο και για την αρχή της ε, εταιρικής συνεργασίας. Κάτι το οποίο χάθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα φροντίσουμε λοιπόν η αρχή της ε, εταιρικής συνεργασίας να παραμείνει πλήρως ισχυρή όπως έως τώρα και να μην αποδυναμωθεί. Ευχαριστώ. Thank you, Demato. Ευχαριστούμε, κυρία Μάτο. Ήθελα να επισημάνω ότι στην πραγματικότητα αυτό το 4% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του νέου, του plus, το 4% είναι λίγο. Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι παραπάνω, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Δεν δίνεται λοιπόν και τόσο μεγάλη προσοχή από πλευράς Κομισιόν. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου όσον αφορά τη συγκέντρωση των διαφορών θεματολογιών, το γεγονό ότι η καταπολέμηση τη φτώχεια και η κοινωνική πρόθεση ε, προορίζεται να είναι τουλάχιστον το 25%. Έτσι αναγνωρίζουμε και εμείς και η Κομισιόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια έκτακτη ανάγκη που απαιτεί συντονισμό και αποτελεσματικότητα στην απόκριση. Αν δούμε τα στατιστικά στη χώρα μου, μιλάμε για 5 εκατομμύρια ανθρώπους ε, στην απόλυτη φτώχεια. Το 2016 και 2017 αυξήθηκε η φτώχεια σε θέμα οικογενειών. Ένα εκατομμύριο 788.000 οικογένειες, 5 εκατομμύρια 58.000 άνθρωποι. Ε, όλοι αυτοί ζουν στη φτώχεια. Γι' αυτό σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχει ακόμα ένας κατώτατος μισθός. Ε, ήθελα να ζητήσω και διευκρινήσει από την Κομισιόν όσον αφορά τη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Στην αιτιολογική σκέψη 21 λέει ότι για να ενισχυθεί η ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τα κράτη-μέλη πρέπει να δεσμεύουν επαρκές ποσό από τους δικούς τους πόρους ε, στο κοινωνικό ταμείο βασί συστατικών ανα... Ε, συστα... Ε, συστάσεων αναχώρα για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων μέσω πολυετών επενδύσεων που εντάσσονται στο κοινωνικό ταμείο. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 7 και στο άρθρο 11 η διαταξή που περιλαμβάνεται στο Common Provision Regulation ε, συνοδεύεται από το άρθρο 15 των κοινών διατάξεων όπου λέγεται ότι η Κομισιόν δεν θα έχει μόνο την εξουσία να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις ε, συστάσεις αναχώρα αλλά θα μπορούσε μονομερός να αναστείλει πληρωμές ε, εξ ολοκλήρου ή εν μέρη του προγράμματος και θα ήθελα ειλικρινά κάποιες εξηγήσει Τι εννοεί η Κομισιόν με συστάσεις σημαντικές αναχώρα. Τι σημαίνει με το κατάλληλο ποσό δεσμευμένο για τις συστάσεις. Συστάσεις που όπως ξέρουμε όλοι αφορούν συγκεκριμένες προτάσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στη χώρα μου, στην Ιταλία, ορισμένε συστάσει αναχώρα για το 2018 είναι για παράδειγμα σχετικέ με την μείωση των ε, ε, συντάξεων γύρατος ε, ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για να μπορέσουν να δαπανηθούν τα χρήματα άλλο. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κανένα άλλο να θέλει να σχολιάσει. Αυτά ήταν λοιπόν τα σχόλια τις εισηγήτρες πρώτα απ' όλα, τη συντάκτριάς μα, των σχεδόν εισηγητών και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε και εσείς το λόγο. Η κυρία Ντεμόντι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την ε, συντάκτρια της νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ και τους σκιώδες συζητητές για τα σχόλιά τους όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ESF+. Θα κάνουμε διάφορες τεχνικού χαρακτήρα παρουσιάσεις και στην Επιτροπή ΕΜΠΛΟ και σε άλλους ευρωβουλευτές ε, δηλαδή και να ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί. Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για διευκρινήσεις τεχνικού χαρακτήρα, ευχαρίστως. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πρόταση με στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη συγχώνευση διαφόρων προγραμμάτων, αλλά όχι μόνο. Και πολύ πιθανόν να χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις ένα μήνυμα τώρα όσον αφορά τη σύνδεση του ESF με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πράγματι, η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η σχέση αυτή να γίνει ακόμα πιο στενή. Όμως, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα θετικά και τους στόχους της διαδικασίας. Δηλαδή, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση, χωρίς όμως να πλήξουμε τι επενδυτικές πολιτικές, αλλά ούτε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, που στο κάτω-κάτω έχει τη δικιά του διαδικασία, συζητήσεις με τις χώρες μέλη κτλ. Και γιατί δεν βάλαμε συγκεκριμένο ποσοστό για τους κατάλληλους πόρους που πάνε στις χώρες από τις ειδικέ συστάσεις. Θελήσαμε να αφήσουμε περιθώριο για συζητήσεις στην διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων στη συζήτηση με τις χώρες μέλη, να δούμε δηλαδή τελικά ε, τι πόροι θα επενδυθούν και σε τι τομεί προτεραιότητα. Αλλιώ θα ήταν σαν να βάζαμε στενό κορσέ στι χώρε μέλη, αν βάζαμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Υπάρχουν ε, βέβαια στοιχεία που παραμένουν ανοιχτά και μπορούν να συζητηθούν στι διαπραγματεύσει και στο Συμβούλιο από τις χώρες μέλη, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ε, ενθουσιασμό σας και να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Σημαντικό αυτό που λέτε, ότι είσαστε ανοιχτοί για παρετέρω συνεργασία και επιπλέον πληροφορίες αν χρειάζονται. Κύριε Παρακαλώ, αργήσατε. Ναι, ναι, ήμουνα έξω. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ακόμα σκεφτόμουν τις απαντήσεις που πήραμε από την Αυστριακή Προεδρία. Τέλος πάντων, επανήλθα όμως, ε, για να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτά που ακούω, και είναι και κάτι που και εμένα με απασχολεί, όχι τόσο το θέμα της σχέσης των χωρών ε, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εντάξει, τα κοινωνικά πρέπει κανείς να κάνει πολλές αλλαγές, αλλά εμένα με απασχολεί το επίπεδο. Και παίρνω, σαν παράδειγμα, τη χώρα μου. Το κοινωνικό ταμείο το έχουμε πάει στον Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Έτσι, από εκεί το διευθύνουν. και υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο πήγε στις περιφέρειες. Και προσπαθήσαμε να έχουμε τις δύο πλευρές του νομίσματος. Και μετά στη Σόφια που έγινε συζήτηση στη διάσκεψη, είχαμε την αίσθηση από αυτά που ακούσαμε ότι η σχέση αυτή και η διάρθρωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη, σε περισσότερη κεντρική ε, δίκηση. Δηλαδή είναι παραπάνω χρήματα για την κεντρική δίκηση. Βέβαια, μας ενδιαφέρει το πόσο η σκοπιμότητα πρώτα απ' όλα και θα ήθελα να το διευκρινίσω περισσότερο. Γιατί αν δεν γίνεται περιφερειακά είναι κρίμα, γιατί ο κόσμος τι σκέφτεται. Θα πάμε στο Υπουργείο Απασχόλησης και από εκεί θα πάρω κάτι για την από την Ευρώπη. Όχι, είναι κάτι που πρέπει να είναι κοντά ε, στον κόσμο δεν πρέπει να είναι στο Υπουργείο Απασχόληση της Ολλανδία. Όχι, πρέπει να είναι στην περιφέρεια για να είναι πιο κοντά στο κόσμο και να το καταλαβαίνει ο κόσμος καλύτερα. Εντάξει, άρα παράδειγμα προ αποφυγή αυτό της χώρας σας. Ναι. Η κυρία Μπρέσο, παρακαλώ. Συμφωνώ με τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Είναι ανησυχητικό το θέμα. Θα μιλήσω τελικά τώρα. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Πράγματι. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ότι ενώ υπάρχει η ανάγκη με την οποία πιστεύω συμφωνούμε όλοι ε, να συντονίσουμε τις ε, περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές ε, και τις εργασιακές πολιτικές και πολιτικές κατάρτισης σε συνάρτηση με τις ε, ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξωμένου και τις συστάσεις αναχώρα. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει κίνδυνος επανεθνικοποίησης των ταμείων και να χωριστεί το κοινωνικό ταμείο, να αποχωριστεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό είναι η κύρια ανησυχία. Θα το δείτε και στις τροπολογίες, ε, όπου εμείς υπενθυμίζουμε διαρκώς την εξή αρχή ότι οι πολιτικές αυτές μπορούν να καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο και σίγουρα πρέπει διότι αποτελούν το γενικό πλαίσιο. Στη συνέχεια όμως η συγκεκριμένη διαχείριση των ταμείων και οι συγκεκριμένες πολιτικές ε, δεν μπορούν παρά να είναι περιφερειοποιημένες. Ειδικότερα στις μεγάλες χώρες είναι αδιανόητο να φανταστούμε να έχουμε τις ίδιες πολιτικές εργασίας παντού. Θα ήταν πολύ δύσκολο τις εποχές ακριβώς που αυξάνονται οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών εμείς να επανεθνικοποιούμε τους πόρους. Αυτή η ανησυχία ε, γίνεται αμέσως ε, προφανής ε, όταν διαβάζει κανείς το κείμενο. Είναι και μια ανησυχία που εμείς απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε κάποιες διαβεβαιώσεις από μέρους της. Εγώ το είχα πει πολύ προσεκτικά, αλλά αυτή είναι η κύρια μας ανησυχία το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ε, να λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις της συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το πώς η κάθε χώρα μπορεί να επιδιώκει αναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές ε, ε, κοινωνικής ένταξης ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ε, επικέντρωση στην ισχυρή αύξηση, όπως είπε και η συνάδελφος κυρία Μάτο, αύξηση λοιπόν της στόχης στις διαφορε χώρε. Αυτό όμως δεν μπορεί να σημαίνει επανεθνικοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Κοινωνικής Ανάπτυξης ε, που είναι το άλλο σκέλος των περιφερειακών πολιτικών όπως είπα χώρες στο οποίο οι πολιτικές ε, περιφερειακής ανάπτυξης που είναι ένας από τους στόχους της πολιτικής σύγκλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Είναι αδιανόητο για παράδειγμα να έχουμε καινοτόμε πολιτικές σε διάφορους τομείς εάν δεν υπάρξει προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού των ανθρώπων. Οι πολιτικές ε, αποσκοπούν ε, να χρησιμεύουν στου ανθρώπου ε, πρώτα απ' όλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπτύξουν αυτέ τι νέε πολιτικέ, δεν θα χρησιμεύσουν τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα. Διάφοροι συνάδελφοι έκαναν κάποιες παρατηρήσεις λαμβάνουμε υπόψη το ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση παρότι δεν αποτελεί κομμάτι του γενικότερου πακέτου ωστόσο Αναμφίβολα είναι ένα από τα θέματα που συχνά απαιτούν κάποια προσαρμογή των ενεργών πολιτικών εργασίας και προσαρμογή των ενεργών πολιτικών κατάρτισης των ανθρώπων. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Όπως και η ισότητα μεταξύ των φύλων, που δεν νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει. και κάτι άλλο που εγώ για να πω την αλήθεια δεν το υπενθύμισα αλλά το γεγονός ότι με το 10% για τις ε, ειδικέ πολιτικές για τους νέους ε, είναι σημαντικό διότι σε αυτή την περίπτωση εμείς ε, συγχωνεύουμε την εμπειρία του Youth Guarantee και στόχος του να της συγχώνευσης του Youth Guarantee στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ακαδημίο Πλάσσα είναι να αξιοποιηθεί η θετική εμπειρία του Youth Guarantee αλλά να γίνει πιο διαρθρωτική, πιο δομική. Να ενταχθεί πλήρως λοιπόν στον κύριο κόρμο το πολιτικό να μην αποτελεί μια περιφερειακή πολιτική αλλά μια από τις κύριες πολιτικές διότι πλέον από διαρθρωτική άποψη αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα της ανεργίας των νέων ε, εντός ενός ευρύτερου σοβαρού προβλήματος υψηλών επέδρων ενέργειας σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Ε, αλλά ειδικότερα η ανεργία των νέων είναι παντού πιο υψηλή, οπότε είναι ένα πρόβλημα που αφορά συγκεκριμένα τους νέους και θα πρέπει να αποτελέσει δομικό υλικό ε, της πολιτικής ολόκληρου του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Πλάς και όχι μόνο ένα κομματάκι του. Γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά έχει συμπεριληφθεί. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το ξεχάσουμε. Ευχαριστούμε. Εδώ τελειώνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και περιμένουμε το κείμενο το Σεπτέμβριο, έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη προετοιμασία, για την παρουσία σας, όλα. Ωραία, συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη και πάμε πάλι στην ε, επίσκεψή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, τα ακούσαμε αυτό, μας τα είπε ο κύριος Ομερζέ. Είμαστε στην έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Υπάρχουν σχόλια? Εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών. Έχουμε τίποτα στα διάφορα? Όχι. Καλώς. Επόμενη συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο. 3 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ και τους Δερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Τους ευχαριστούμε πραγματικά για τη δουλειά τους. Και εύχομαι σε όλους σας καλές διακοπές. Καλό ηλιόλουστο καλοκαίρι.